Pan Przewodniczący! Witam Państwa e, obecnych na e, kolejnym posiedzeniu. Σας ε, χαιρετίζω καρδιότατα και κυρίως την της σημερινής μας συνεδρίασης. Ευρωπαϊκή Ράτζε το πρώτο σημείο της ημερησίας διάταξη είναι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τη 16 η και 17 η Δεκεμβρίου. Δηλώσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη Επιτροπή. Σύμφωνα με τις ειδήσει τη Λισαβόνας θα κάνει καταρχήν μια παρουσίαση ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Χερμαν Van θα κάνει μια παρουσίαση και σα καλωσορίζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Uh, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχηθώ σε όλους ένα ευτυχισμένο νέο έτος. Σας το εύχομαι προσωπικά για σας κύριε Πρόεδρε, αλλά και για ολόκληρη την Ένωση σε αυτούς τους κρίσιμους